République tunisienne. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τινησίας. Meine sehr geehrten Damen und Herren. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι μεγάλη τιμή για μας να σας παρουσιάσω εδώ, να καλωσορίσω τον πρόεδρο της Τινησιακής Δημοκρατίας, Μονσέφ Μαρζούκη, στο Στρασβούργο. Καλώς ήρθατε, κύριε πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, ενώ ήρθατε εδώ, Πενδύει ταυτόχρονα η χώρα σας τον ηγέτη του λαϊκού μετόπου Σοκέ Μπελαΐτ, ο οποίος σήμερα το πρωί θανατώθηκε, δολοφονήθηκε με φρικιαστικό τρόπο. Ε, καταδικάζουμε βεβαίως αυτή την επίθεση εντόνως. Γνωρίζουμε ότι οι τυνησιακές αρχές θα πράξουν ό,τι περνάει από τα χέρια του και θα λάβουν τα αναγκαία μέτρα ούτω ώστε να προσαγάγουν τους υπεύθυνους ενώπιον της δικαιοσύνη. Ένα τέτοιο έγκλημα δεν θα πρέπει να παραμείνει ατιμόρυτο. Θα ήθελα να συλληπιθώ την οικογένεια του κυρίου Μπελαΐντ και τον τυνησιακό λαό σε αυτή τη δύσκολη ώρα βρισκόμαστε στο πλευρό σας και απευθύνω μία έκκληση προς όλους τους πολίτες της Τινησίας να υψώσουν το ανάστημά τους και να προσχωρήσουν στο πνεύμα της δημοκρατίας ούτως ώστε να κατησχίσει το πνεύμα της συμφιλίωσης που οδήγησε στις 12 Ιανουαρίου 2011 στην απελευθέρωση της χώρας. Ούτως το πνεύμα αυτό της συμφιλίωσης να παραμείνει ζωντανό. Κύριε Πρόεδρε, στο δικό σας πρόσωπο αγκαλιάζουμε με ανοιχτά, δεχόμαστε μάλλον με ανοιχτές αγκάλες τον εκπρόσωπο ενός θαραλέου λαού. Η επιτυχία του οδήγησε πριν από δύο χρόνια ε, στην, ε, στον τερματισμό της εξουσίας, μιας διαφερμένης εξουσίας. Κύριε Πρόεδρε, εδώ ε, στην αίθουσα της Ολομέλειας, της Ολομέλειας παρακαλώ να μνημονεύσετε και το λαό της Τινησίας που πλήρωσαν ε, με τη ζωή τους τη μια αξιοπρεπή και ελεύθερη ζωή. Τέλος, ε, κυρίες και κύριοι, καλωσορίζουμε μαζί με τον πρόεδρο της ε, Τινησίας εδώ, σε αυτή την πόλη, έναν άνθρωπο ο οποίος ε, ήταν γιατρός και εξόριστος, γιατί 15 χρόνια έζησε εδώ στο Στρασβούργο, αφιερώνοντας ε, τις προσπάθειές του για το, στο καλό των ασθενών του, αγωνιζόμενος για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, ο κύριος Πρόεδρος ε, μου είπε ότι ως πολίτης του Στρασβούργου συνέβαλε στην δημιουργία του παλαιού ή μάλλον παρέστη ως μάρτυρας στην δημιουργία του, του παλαιού του Κοινοβουλίου και του καινούριου κτηρίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, και για μένα είναι πραγματικά μια στιγμή μεγάλη συγκίνηση Σαν κάποιος ο οποίος έζησε επί 23 χρόνια εξόριστος κοντά σε αυτό το κτίριο το οποίο πάντοτε υπήρξε το σύμβολο για την ελπίδα ότι κάποια μέρα θα φωτίσει η ελπίδα της ε, της ελευθερίας στη χώρα μου. Ε, κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι και για μας η στιγμή αυτή είναι συναισθηματικά φορτισμένη. Το γεγονός ότι μπορούμε να σας καλωσορίσουμε εδώ. Ο λαός σας ε, τερμάτισε την αυθαιρεσία το θέρτο καθεστώ και έθεσε θεμέλια ενό κράτους δικαίου. Ο δρόμος αυτός ε, ήταν ε, μακρύ ε, και δύσκολος και παραμένει επώδυνος. Ωστόσο, παραμένω πεπισμένος ότι για την χώρα σα δεν θα υπάρξει καμία οπισθοχώρηση, αλλά θα συνεχίσετε στον δρόμο της δημοκρατίας. Εγώ το Δεκέμβριο ήμουν προσκεκλημένος σας στην Τίνιδα και για πρώτη φορά πήγα τότε στην Κινησία και θα πρέπει να ομολογήσω ότι πραγματικά αισθάνθηκα κάπως αμήχανος τότε γιατί δεν, δεν ήξερα πώς ε, ε παρουσιάζεται μια χώρα που βρίσκεται σε μια διαδικασία μετάβασης αλλά θα πρέπει να σας πω ότι το θάρρος το, και το κουράγιο των ε, πολιτών πραγματικά με συγκλώνησαν. Ε, μου εξηγήσατε ειλικρινά ότι ο ρόλος σας ως Προέδρου είναι να δώστε το αίσθημα ε, εμπιστοσύνη προς όλους τους πολίτες, σε εκείνους που αγωνίζονται για την βελτίωση της ε, δημοκρατίας. Θέλετε να δώσετε σε όλους αυτούς μια ελπίδα. Θεωρείτε ότι αυτό είναι το έργο σας και το μέλημά σας κύριε Πρόεδρε. Αλλά για να το επιτελέσει αυτό ένας πρόεδρος χρειάζεται μια υποστήριξη. Και για να λάβετε αυτή την υποστήριξη ήρθατε εδώ σε αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα την πάρετε, θα την έχετε σίγουρα. Καλώς ήρθατε κύριε Πρόεδρε και έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, αγαπητοί φίλοι, από το 1996 στο 2001 η δικτατορία μου είχε απαγορεύσει να καταλήψω την Τινησία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απάντησε σε αυτό με αυτό το έγγραφο το οποίο σας δείχνω. Το διαβατήριο της ελευθερίας το οποίο διδόθηκε στην μικρή κόρη μου εδώ ακριβώς αυτό το χώρο του 2000. Είναι ένα συμβαλικό διαβατήριο το οποίο υπογράφουν η Ελέν Φλότρε, ο Ζαν Μισελ Ροκάρ, Αστρίτ Τόρς, Τζαν Φράνκο Ντελάλμπα, Ντανιέλ Κονμπεντίτ, Ντανιέλ Ντικάρμ, Ζωζέ Μαρία Μεντιλούτσε, Αλέν Λιπίτς, Φοντέ Σίλα, Αλή Ματιέρη Μπουμεντιέν, Σεσίλια Μάλμστρομ, Μαρία Αρλέτ Καρλώτη, Φρανσουάς Γκροστέτ και Φρανσουά Ζιμερέ. Αν μου επιτρέπετε θα ήθελα να εκφράσω σε όλους ε, αυτούς ε, τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη και για όλους ουσιαστικά, διερμηνεύοντας ε, την ευγνωμοσύνη και των άλλων, για όλους τους ε, Άραβες και την ίσως δημοκράτες ε, που πάντοτε βρήκαν σε, αυτή την, σε αυτό το χώρο εδώ που εκπροσωπείται την πιο απερίφραστη υποστήριξη. Κυρίε και κύριοι, στα τέλη δεκαετία του 1990 είχα γράψει ότι αν ο 18ο αιώνα ήταν ο αιώνα τη Γαλλική και Αμερικανική Επανάσταση, ο αιωνα τη γαλλικη και αμερικανικη επανασταση ο 20 τη Κινέζικη και Ρωσική επανάσταση, Ο 21 ο αιωνα θα είναι ο αιώνα τη Αραβική Επανάσταση. και αυτό δεν το διάβασα στο φλιτζάνι του καφέ, αλλά ξεφύλλοντα τι σελίδε τη ιστορία. Ε, τα μεγάλα έθνη ούτε αυτοκτονούν ούτε πεθαίνουν. Και όταν όλα φαίνονται χαμένα, τελικά ανασύρουν από τα βάθη την ενέργεια και ξανασηκώνονται. Όσο πιο μεγάλο ο Γολγοθά ε, και πιο βαθιά η πτώση, τόσο πιο μεγάλη ενέργεια που θα τους βγάλει από αυτή την τρύπα και αυτό είδαμε και στις αραβικές επαναστάσεις. Είναι ένα είδος ε, ε επαναλαμβανόμενης, ε, ε επαναλαμβανόμενη γεγονότος στην ιστορία. Το θέμα είναι τελικά ε, για όλους τους Ευρωπαίους αν αυτές οι επαναστάσεις για μας είναι καλό ή κακό, αν είναι ευκαιρία ή κίνδυνος. Για να καταλάβουμε όμως όλα αυτά θα πρέπει να έχουμε και μια ελάχιστη δόση ενσυναίσθησης γιατί αλλιώς ε, ούτε βλέπουμε ούτε καταλαβαίνουμε. Και δεν ζητώ απλά την προσοχή σας λοιπόν, ζητώ την εν σα, σας, γιατί δεν θα μπορέσουμε ούτε να επικοινωνήσουμε ούτε να συναντηθούμε. Ναι, οι αραβικές επαναστάσεις μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στην Ευρώπη. Ήδη βλέπουμε τα βασικά από αυτά. Υπάρχει ο κίνδυνος ότι θα προκύψουν ταραχές, ίσως και εμφύλοι πολέμοι όπως βλέπουμε στη Συρία. Με όλα αυτά τα αρνητικά μπορεί να έχουν για την ασφάλεια στην Ευρώπη. Το δεύτερο κίνδυνο, τον είδαμε μετά την τόση δικτατορία στην Τινησία, είναι ότι οι νέοι μα που βλέπουν να καταραίει το, ο μηχανισμό ασφάλεια και ξέροντα και τι οικονομικέ δυσκολίε, ε, μπήκαν ε, στα πλοία και ήρθαν ε, στι ακτέ τη Ευρώπη, βλέποντα εκδό την ελπίδα. Επίση, έχουμε μια άλλη τρίτη απειλή, τον Ισλαμικό εξτρεμισμό, τον τζιχαντιστικό σαλαφισμό, όπω τον λέμε, που θα μπορούσε να πάρει νέα όθηση. Επίσης, ε, στην περίπτωση Αλκάιντα έχουμε ε, μια παγκόσμια απειλή, αλλά έχουμε και μια περιφερειακή απειλή, όπως το Βόρειο ε, Μαλί, που είδαμε ότι ξεκίνησε και λόγω αυτής η Γαλλική Επανάσταση. Πρόκειται για πραγματικά εθνική απειλή σε όλες τις χώρες της Αραβικής Άνοιξης. Αλλά το σημαντικότερο είναι αυτό και όχι η συνένοχοι του παλαιού καθεστώτος και η Δημοκρατική Επανάσταση έκοψε τα φτερά αυτού, αυτών. Κυρίε και κύριοι, πρέπει να δούμε και μισογεμάτο το ποτήρι, γιατί πραγματικά δεν πρέπει να φοβόμαστε τι αραβικέ επαναστάσει. Δεν είναι εθνικιστικέ ούτε ξενοφοβικέ. Όταν ξεκίνησαν, δεν ακούσαμε ε, ε, συνθήματα κατά τη Δύση, κατά του Ισραήλ. Η ελευθερία ε, ουσιαστικά είναι απέναντι σε μια διεφθαρμένη βία δικτατορία. Είχαμε πρόσφατα κάποιε βίες διαδηλώσεις κατά των δυτικών ε, πρεσβειών λόγω ενός ε, βίντεο ισλαμόφοβου, αλλά μόνο ελάχιστοι ήταν αυτοί οι οποίοι το υποστήριξαν αυτές τις αντιδράσεις. Οι περισσότεροι ήταν κατά και πραγματικά δεν πρέπει κανείς να φοβάται τις αραβικές επαναστάσεις γιατί πρώτα απ' όλα κυρίως είναι κοινωνικές. Αγωνίζονται δηλαδή για τα κοινωνικά οικονομικά δικαιώματα για τα οποία αγωνίστηκατε κι εσείς, τις δικές σας, είτε επαναστάσεις, είτε ε, ειρηνικές, είτε και τώρα δεν θα πρέπει να φοβόμαστε τις αραβικές επαναστάσεις γιατί είναι και δημοκρατικές. Σίγουρα υπήρξαν εκλογικές νίκες στην Ισία, τη Λιβύη, την Αίγυπτο. Ουσιαστικά και από τη δημοκρατία προέκυψε η άνοδος Ισλαμιστών και δεν πρέπει να θεωρούμε ότι οι Ισλαμιστές είναι αυτοί οι οποίοι έχουν θριαμβεύσει ή ότι μπορούν στη συνέχεια να διαστρεβλώσουν τα πράγματα. Η δημοκρατία παραμένει, παραμένει στον κόσμο. Ουσιαστικά πρέπει να πούμε ότι είναι δημοκράτες και οι Ισλαμιστές. Τώρα θα δούμε αν είναι ε, ειλικρινείς, θα το δείξει ο καιρός, αλλά θα πρέπει να ξαναμάθουν ε, να παίζουν σύμφωνα με τους κανόνες για να μην έχουμε μια θρησκευτική δικτατορία, την οποία όμως και αυτοί οι Άραβες θα την ε, πατάξουν. Σε ό,τι αφορά σε ό,τι αφορά αυτούς οι οποίοι ήδη μιλούν ε, για τον Ισλαμικό χειμώνα μετά την Αραβική Άνοιξη, φαίνεται ότι δεν βλέπουν ότι χρειάστηκε πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες και σε άλλους λαούς για να μπορέσουν να εξορροπήσουν μετά από μια επανάσταση. Βέβαια ε, δεν έχει τίποτα κρυθεί ακόμη σε ό,τι αφορά το τι θα γίνει με αυτέ τι επαναστάσει. Για την Τινησία, τη χώρα μου που ξέρω καλύτερα, μπορώ να σα πω ότι είμαστε περήφανοι για αυτή την επανάσταση που δεν στήχησε παρά ελάχιστα σε ό,τι αφορά ε, τι ανθρώπινε ζωέ και πραγματικά βλέπω με πάρα πολύ μεγάλο πόνο ε, το γολγοθά που βιώνουν ε, οι Σύροι που πληρώνουν πολύ ακριβά την ελευθερία τους, αλλά έχουν και την στήριξη στα ανθρωπιστική την πολιτική όλων των ελεύθερων λαών. Εμείς έχουμε συγκροτήσει μια κυβέρνηση συνασπισμού, ε, έχουμε δύο εξυγχρονιστικές και άλλα παραδοσιακές ε, συνιστώσεις, κοσμικούς αλλά και μετριοπαθείς Ισλαμιστές. Είναι μια κυβέρνηση που λειτουργεί, ε, ξαναορθώνει, στην στα πόδια το κράτος που είχε πάψει να υπάρχει το 2011. Έχουμε μεγάλη ανάπτυξη, συν 3,5% το 2012. Ε, βέβαια έχουμε και κάποια προβλήματα γιατί υπάρχουν πολιτικά και προσωπικά προβλήματα αλλά νομίζω ότι θα πρέπει έτσι να προχωρήσουμε τις επόμενες εκλογές. Ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα αστικό δημοκρατικό κράτος, μια πλουραλιστική κοινωνία. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά έχουν δυσκολίες ε, αλλά ε, σύντομα θα τα καταφέρουμε και ελπίζω να έχουμε και ένα κείμενο το οποίο θα ε, είναι έτοιμο μέσα σε δύο-τρει μήνε. Ξέρετε ότι μέσα σε δύο χρόνια δεν μπορεί να αλλάξουν νοοτροπίε 50 ετών. Βέβαια, θέλουμε να διαφυλάξουμε τον τρόπο ζωή ε, τη ε, σύγχρονη νησίας και να αυξήσουμε το βιωτικό επίπεδο και των φτωχών ξεχασμένων ε, την ίσιον. Έχουμε όμως τεράστιες κοινωνικο-οικονομικές προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε. Είναι βαριά κληρονομιά της δικτατορίας που ήταν πολύ καλά συγκαλυμμένα όλα αυτά εδώ και 20 χρόνια. Θέλουμε όμως να συνεχίσουμε τη στρατηγική μας ε, ε, γιατί μπορεί να μην βλέπουν κάποιοι ιδεολόγοι την πολυπλοκότητα και τη δυναμική των πολιτικών δρομένων. Εμείς όμως θέλουμε να ενισχύσουμε τη μετριοπαθή συνιστόσα, την Ισλαμιστική και συγχρόνως να ε, σεβαστούμε βέβαια και τη, τη, τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και την κοινωνικο-οικονομική και πολιτισμική ανάπτυξη. Αυτό το ρεύμα, δηλαδή το αντίστοιχο της δικής σας ακροδεξιά, θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο αυτό το μοντέλο της ε, κοινωνίας που βασίζεται στην αραβομουσουλμανική κληρονομιά και στρέφεται προς το μέλλον. Δεν θα αφήσουμε να μπουν σε κίνδυνο τα κεκτημένα για τη γυναίκα και τα ανθρώπινα δικαιώματα, σχέση μας με τη Δύση που θέλουμε να συνεχιστεί να είναι ειρηνική, φιλική και να βασίζεται στον αλληλοσεβασμό. Κυρίε και κύριοι, βέβαια υπάρχουν εμπόδια, πάρα πολλά εμπόδια σε αυτό το δρόμο, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί ε, που είναι εχθρικοί σε αυτή την ειρηνική επανάσταση και θέλουν να αποτύχει. Βλέπουμε φραστική βία. Ε, στρέφονται οι μουσουλμάνοι κατά των μουσουλμάνων. Και σήμερα είχαμε αυτή τη φρικτή δολοφονία ενό προηγέτη αντιπολίτευση, ενό πολιτιστικού ηγέτη, τον οποίο γνωρίζω πολύ καλά, που για μένα ήταν φίλο εδώ και καιρό. Πραγματικά σήμερα ο Τσόκρι Μπελαΐντ ε, δολοφονείται και είναι σαν ε, να γίνεται επίτηδες. Ήξεραν ότι θα έρθω εδώ σήμερα. Αυτό το μήνυμα δεν θα το ε, λάβουμε. Αυτή την επιστολή δεν θα την παραλάβουμε. Το μήνυμα αυτό δεν πρόκειται να το δεχθούμε και θα συνεχίσουμε για να αποκαλύψουμε, για να βγάλουμε τα πρόσωπα όλων αυτών στο φως. και θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε την πολιτική μα. Η διαδικασία αυτή εκδημοκρατισμού του κράτου και τη κοινωνία, τη δημιουργία μια βιώσιμη ε, δίκαιη ανάπτυξη, φαίνεται, ε, όπω καταλαβαίνετε, πιο δύσκολη, πιο πολύπλοκη, αλλά και πιο μακροχρόνια διαδικασία. Προχωρά όμω. Ε, πολλοί παράγοντε αποφασίσουν για τη μοίρα αυτή τη επανάσταση και όλων των άλλων στι αραβικέ χώρε. Η αποφασιστικότητα των λαών, η η αποθάρρυνσή του, η σοφροσύνη του, η τρέλα του, αυτό το φαινόμενο τη πεταλούδα που είναι δύσκολο κανεί να το ελέγξει ή να το ε, εντοπίσει αλλά μπορείτε να στοιχηματίσετε υπέρ της Τινησίας που είναι πραγματικά ένα εργαστήριο ε, μιας μεγάλης μετάβασης που θα πετύχει πιστεύουμε. Κυρίες και κύριοι έχουμε υποφέρει πολύ στην Τινησία γιατί έλειπε ε, ένα εθνικό κράτος δικαίου αλλά έλειπε αυτό και στο διεθνές επίπεδο. Μετά τις ε, προεδρικές ε, εκλογές που οργάνωνε ο δικτάτορας και κέρδιζε με μόνιμο αποτέλεσμα 99% εμείς οι δημοκράτες, οι αγωνιστές των ευρωπαϊκών δικαιωμάτων το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν να στήσουμε την ακύρωση των αφευμένων αυτών, αλλά δεν υπήρχε ούτε συνταγματική, συνταγματικό εθνικό δικαστήριο, ούτε διεθνέ. Εξού και ήρθε αυτή η ιδέα να έχουμε αυτό τον υπερεθνικό φορέα που θα αποφασίζει με βάση την Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρώπινα Δικαιώματα ε, το κατά πόσον ε, συμφωνούν και συνάδουν ε, οι εκλογέ με τις διεθνείς συνθήκες. Και αυτός ο οργανισμός πήρε, την, πήρε το πράσινο φως από την Αφρικανική Ένωση της Αμπέμπα την προηγούμενη εβδομάδα και έτσι το κράτος δικαίου παγκόσμια θα συνεχίσει να προχωρά και η δημοκρατία θα συνεχίσει να ενισχύεται. Κυρίες και κύριοι, οπωσδήποτε θα πρέπει να βασιστούμε στις δυνάμεις μας, αλλά θα θέλαμε να μπορούμε να στηριχτούμε και στην Ευρώπη. Για πρώτη φορά στην κοινή μας ε, ιστορία και την κοινή μας πορεία ταυτίζονται ε, οι ε, απόψεις μας. Έχουμε κοινά συμφέροντα. Μέσω πρόθεσμα όμως είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να επιτύχουμε την εξυγίαση της οικονομίας μας, έτσι ώστε να εξηγιάνουμε ταυτόχρονα και την αναδυόμενη δημοκρατία μας. Ευχαριστούμε και τη Γερμανία, η οποία δέχτηκε να αναλάβει αναλάβει ένα μέρος του χρέους μας, 60 εκατομμυρίων ε, ευρώ ε, μέσα σε προγράμματα ανάπτυξης και ελπίζουμε ότι και οι άλλοι εταίροι, κυρίως ε, η Γαλλία, θα κάνουν το ίδιο. Κυρίες και κύριοι, πέρα από αυτά τα οικονομικά στοιχεία υπάρχουν στις σχέσεις μεταξύ των δύο κόσμων μας και πράγματα πιο ουσιώδη. Ε, οι ε, αστρονόμοι ε, ασχολούνται με, τις, με τους γαλαξίες και εμείς μπορούμε να ταυτοποιήσουμε πολιτισμούς και ομάδες πολιτισμών. Μην ξεχνούμε ότι Μαχρέμπε σημαίνει στα αραβικά Δύση και επομένως με αυτή την έννοια εμείς που είμαστε στην Δύση είμαστε όμως ε, και ε, η Δύση που μοιράζεται την, ε, τον Νότο μαζί με τους βόρειου και ξέρουμε ότι η Δύση οφείλει, οφείλει κάποια πράγματα στον άραβο-μουσουλμανικό πολιτισμό. Γνωρίζουμε επίσης ότι ο εξυγχρονισμό της άραβο-μουσουλμανικής κουλτούρας έχει εν μέρη μάλλον οφείλεται στην Ευρώπη η οποία δημιούργησε και μεγαλούργησε πολλά βασιζόμενο σε αυτόν τον πολιτισμό. Ε, η ιστορία των Αράβων που είναι τριών 300 ε, εκατομμυρίων ετών ε, είναι μεγάλη. Εκεί βασίζονται οι ευρωπαϊκές γλώσσες και αυτό είναι το κληροδότημα που έχουμε δώσει στις επόμενες γενιές. Η ευρωπαϊκή επιρροή στον αραβικό κόσμο ε, είναι επίσης ιδεολογική και αυτό δεν είναι πρόσφατο. Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα ε, η Αίγυπτο το Ιράκ και η ε, Λιβύη είδαν τον εαυτό του στο ρόλο τη Προύσα, του Νασέρ, του Σαντάμ και του Κατάφη που ήθελαν να γίνουν οι νέοι Άραβες Μπίσμαρκ. Αυτό το μοντέλο Αραβική Ενότητα που βασίζεται στο, χάρισμα του ηγέτη και, και στα όπλα έχει πτωχεύσει πλέον και ευτυχώ Δυστυχώς ε, σήμερα αυτό που θέλουμε είναι μια μεγάλη ένωση του Μαχρέμπ ε, επί τη βάση του μοντέλου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μας γοητεύει γιατί πραγματικά κατάφερε κάτι θαυματουργό, δηλαδή την γαλλογερμανική ανακοχή και η ύπαρξη ενός τέτοιου θαύματος δείχνει ότι είναι δυνατόν να κάνουμε κάτι τέτοιο και εμείς, έστω και αν τα θαύματα δεν γίνονται κάθε μέρα. Εμείς θέλουμε να ζητήσουμε σε όλους και στους συναδέλφους μας από το Ισραήλ ε, απέναντι σε αυτό το μπλοκάρισμα το οποίο βασίζεται ε, σε υφιστάμενες απειλές αλλά και σε μελλοντικές απειλές ε, να μπορέσει να καταλάβει πώς πρέπει να κινηθεί στο μέλλον. Θέλουμε να τους ζητήσετε να ελευθερώσουν και τον Μαρουάν Μπαρχουτή και να τον αφήσουν να επιστρέψει στην την Ισία ε, για να μπορέσει να ξαναβρει την υγεία του που έχει καταστραφεί μετά από 10 χρόνια ε, στην απομόνωση. Κυρίε και κύριοι, ξεκίνησα με ε, μια προσωπική ενθύμηση. Επιτρέψτε να τελειώσω με κάτι αντίστοιχο. Στο Στρασβούργο έκανα τις σπουδέ μου. Εδώ έμαθα τη δουλειά μου. Είναι η χώρα η οποία και η πόλη μάλλον, οι πολίτες της οποίας χάραξαν μέσα μου την έννοια της εργασίας, της μετριοπάθεια, ε, τη υπιότητας. Ε, εδώ γεννήθηκαν και οι, οι, οι ε, κόρες μου. Ε, ξεκίνησα στην αρχή της δεκαετίας του 70 σαν νέος ε, γιατρός ε, και ζήτησα από έναν καθηγητή να μου δώσει ένα θέμα για την διπλωματική μου εργασία. Μου πρότεινε ένα θέμα που αφορούσε τις, τα ανθρώπινα πειράματα στην ιατρική. Δεν το δέχτηκα γιατί με ενδιέφερε τόσο πολύ, αλλά γιατί την έκανα αυτή τη διατριβή με τον Μάρκ Κλέιν είναι και ήξερα ότι ε, ως Εβραίος είχε περάσει από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και ως ε, γιατρός ε, είχε κάνει πάρα πολλά τέτοιου είδους ε, ε, πειράματα. Η προετοιμασία αυτής της διατριβής ήταν τελικά ένα ταξίδι ε, στην Φρίκη. Ο Μάρκ Κλάιν δεν νομίζω ότι είχε καταλάβει εκείνη την εποχή τον αντίκτυπο που θα είχε σε αυτόν τον νεαρό γιατρό που του ζήτησε τη διατριβή, ούτε ότι θα είχε καταλάβει τους μυστικούς δρόμους που μου άνοιγε και τους νέους κόσμους που μου άνοιγε. Ε, εγώ τότε ε, δεν μπορούσα και εγώ ο ίδιος και σίγουρα ούτε και ο Μαρκ Κλάιν να κατανοήσουμε ε, πώς θα εξελίσσονται τα πράγματα. Αλλά σήμερα βλέπω ότι έχω επιτύχει κάποιες νίκες και ακριβώς αυτή η τελευταία μου νίκη μου επιτρέπει να είμαι εδώ σήμερα σε αυτό το κέντρο της δημοκρατίας, της ειρήνης και της αδελφότητας μεταξύ των λαών που μου δίνει την δυνατότητα να πάρω το λόγο σήμερα εξ ονόματος ενός λαού ελεύθερου. και τη σημερινή μου παρουσία θα ήθελα να την αφιερώσω σε αυτό το ε, λαό. Θα ήθελα με την ίδια ευκαιρία ε, να χαιρετήσω το Στρασβούργο, την Αλζατία, την ε, Φιλία και την Ευρωαραβική ε, Θρησκεία. Ασαλέμ αλέκουμ και η ειρήνη να είναι μαζί σας. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτα στα λόγια του κυρίου Προέδρου και στα δικά σας χειροκροτήματα. Παρ' όλα αυτά, συμφώνησα με τον Πρόεδρο γιατί ε, έλαβα πάρα, πολλά αιτήματα από τους βουλευτές. Το σώμα αυτό, ε, τιμώντας τα θύματα να κάνουμε ένα ενός λεπτού σιγή στο τέλος αυτής της ε, συνεδρίας. Παρακαλώ να σηκωθείτε από τις θέσεις σας. Ήθελα να σας ε, ευχαριστήσω θερμά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Τινησίας. Νομίζω ότι ήταν μια συγκινητική στιγμή. Ζήτω την Τινησία, ζήτω η ελευθερία, ζήτω η δημοκρατία.